Uh, the sitting is open. I would have an announcement uh, to make uh, in relation Έχουμε μία ανακοίνωση για την Επιτροπή ΙΜΚΟ να ξεκινήσει διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις ε, που ανακοινώθηκε στην αρχή της ε, Ολομέλειας, Δευτέρα 11 Μαρτίου. Δεν έχω λάβει σχετικά με αυτό έτοιμα για ψήφο ε, για ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 69C, παράγραφος 2. Επομένω η Επιτροπή ΙΜΚΟ μπορεί να ξεκινήσει τις ε, διαπραγματεύσει. Πάμε στο πρώτο σημείο τη ημέρησιας διάταξη, το οποίο είναι η δηλώση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι για αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye, δεν υπάρχει επίσης διαδικασία μπλε κάρτας. Θα ήθελα να το δεχτείτε αυτό και αν το δέχεστε, ε, δίνουμε το λόγο στην κυρία Σιώτα για να μας πει την άποψη του Συμβουλίου. Καλημέρα, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι προβουλευτέ. Ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο που με άφησε να εκφράσω την άποψη του Συμβουλίου για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι γνωρίζουμε το μέγεθος και, την, και το επίγον των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή αποδεικνύεται από την πολύ έντονη συζήτηση που έγινε για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η παγκόσμια δράση για την καταπολέμηση α, της κλιματικής αλλαγής δεν αρκεί, όπως αποδεικνύει η έκθεση IPPC. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ηγηθεί στην παγκόσμια προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή υπερασπίζεται τις δεσμεύσεις της και την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και να κρατήσουμε την αύξηση της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου. Επίσης θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις συνεισφορές μας ε, στην προσπάθεια για την, ε, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια μιας πολυμερούς προσπάθειας με τη συμμετοχή και της αεροπορίας και της ναυσιπλοείας. Εμείς είμαστε καθοδόν για να ε, πετύχουμε τους στόχους για την ανανεώσιμη πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα του 2020. Επίσης, έχουμε εντάξει σε νομοθεσία του, τις φιλόδοξες ε, δεσμεύσεις μας για το χρονικό ορίζοντα του 2030, τόσο ώστε να πετύχουμε περιορισμό των εκπομπών τουλάχιστον κατά 40% ε, μέχρι το 2030 σχέση με τις τιμές του 1990. Η ολοκλήρωση του πακέτου για την κλιματική αλλαγή του με ορίζοντα το 2030 ξεκίνησε σε προσπάθειες ε, από το 2015 και τελείωσε με συμφωνίες των δύο συνομοθετών. Οι κανόνες του συστήματος εμπορίας εκπομπών αναθεωρηθήθηκε, ούτω ώστε να πετύχουμε τις μειώσεις των εκπομπών στον, στη βιομηχανία και στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Με μειώσεις εκπομπών μέχρι το 2030 για κάθε κράτος μέλος και για άλλους τομείς όπως ε, τα απόβλητα, ε, ο κατασκευαστικός τομέας και οι μεταφορές. Στο δασοκομικό τομέα ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπομπές στην επικράτειά τους ε, δεν ε, υπερβαίνουν ένα όριο. Επίσης, για την ανάπτυξη των ανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις εκπομπές του, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, ε, καθώς και από το φθοριοποιημένο αέριο, ε, θα επηρεάσει το επίπεδο των επιτυχιών μας. Επίση, οι καλοί κανόνε διακυβέρνηση που συμφωνήθηκαν πρόσφατα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των κρατών μελών, καθώ και τα σχέδια, τα μακροπρόθεσμα για την πολιτική, η υποβολή ε, εκθέσεων ε, για την πρόοδο θα διευκολύνουν την προσπάθεια. Πρέπει να γίνουν περισσότερα όμω για να συνεισφέρουμε στου μακροπρόθεσμου στόχου για τη θερμοκρασία με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική στην ε, Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2020, ζητώντα από όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους εγκαίρως. Με αυτά τα δεδομένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Κομισιόν να παρουσιάσει μία πρόταση για μία στρατηγική για τους ε, μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ε, αρχές του 2019 ε, με βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν. Ε, το Συμβούλιο καλωσορίζει την ανακοίνωση και θεωρεί ότι πρέπει να εστιάσουμε τις συζητήσεις σε διάφορους τρόπους για να πετύχουμε την ουδετερότητα με βάση τους στόχους του Παρισιού. Η ανακοίνωση έχει ήδη συζητηθεί σε συνεδριάσεις υπουργών, των υπουργών υπεύθυνων για το περιβάλλον, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω τομεακές συζητήσεις θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οι συζητήσεις ε, βοήθησαν ε, για να αναγνωριστεί η ανάγκη για δράση και να αναγνωριστεί η σημασία του να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μακροπρόθεσμη στρατηγική μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η συντονισμένη δράση θα πρέπει να φτάσει σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Οι μη κρατικοί εταίροι έχουν σημαντικό ρόλο, οι τοπικές αρχές επίσης έχουν το σημαντικό ρόλο για να εφαρμοστούν φιλόδοξες λύσεις επί τόπου. Η προετοιμασία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ολοκληρωμένου στόχου σε εθνικό επίπεδο που θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης. Να σας υπενθυμίσω ότι η Συμφωνία του Παρισιού αναγνωρίζει ότι η μετάβαση είναι σημαντική ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής λαμβάνονται υπόψη σε περιφέρειες και κοινότητες και δήμους που θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από αυτό. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, για την ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, παρά τα τεράστια προβλήματα. Η μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανθεκτικές οικονομίες έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περαιτέρω θέσεις απασχόλησης, κυρίως στον τομέα των νεώσιμων πηγών ενέργειας, στον κατασκευαστικό τομέα και στην ανακαίνιση κτηρίων. Οι τεχνολογικές ανακαινήσεις θα πρέπει να ενταθούν σε όλους τους τομείς, η έρευνα, η ανάπτυξη. Είναι σημαντικές για να μειώσουν το κόστος των καινοτόμων τεχνολογιών και χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα τη στηρίξει θα πρέπει επίσης να έχουμε και ιδιωτικά εργαλεία για να δώσουμε τα κατάλληλα μηνύματα στην αγορά με κινητοποίηση χρηματοδότησης από διάφορες πηγές. Ε, κινητοποίηση χρηματοδότηση από διάφορες πηγές. Για να μειώσουμε τις εκπομπές με βάση τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σεβαστούμε και να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία του Παρισιού θα, γίνουν, θα πρέπει να γίνουν σε κοινωνικό επίπεδο, σε επιλογές μας, στις επενδύσεις και στην κατανάλωση σημαντικές αλλαγές. Καθώς και στα μοντέλα βεβαίω ε, παραγωγής για την επόμενη δεκαετία. Η Προεδρία θέλει να κάνει περαιτέρω συζητήσεις για την ανακοίνωση της Κομισιόν και σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε ήδη το θέμα στη συνεδρίαση, θα συζητήσει μάλλον στη συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, ούτω ώστε να δώσει καθοδήγηση για την κατεύθυνση και τις πολιτικές προτεραιότητες. Με βάση αυτή την καθοδήγηση το Συμβούλιο θα συνεχίσει να συζητάει με στόχευση και εστίαση, ούτω ώστε να συνεισφέρει την όλη διαδικασία. Το Συμβούλιο επίσης ε, προσβλέπει σε εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, σε διεθνές επίπεδο μέσα στο 2019 που θα είναι μια ευκαιρία για να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να υπάρξει πολιτική βούληση για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, όπως είπε το UFCCC εν ώψη της συνεδρίας που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2019. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συνάδελφοι, όσοι ήρθατε πιο καθυστερημένα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει διαδικασία καστιά και ούτε μπλε κάρτα. Και τώρα ο Επίτροπο Κανιέτε θα πάρει το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα, Επίτροπε, και έχετε το λόγο. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε αυτή την ε, συζήτηση προτεραιότητα για την κλιματική αλλαγή. Οι δικέ σα ε, δικές σας ενέργειες και η προσήλωσή σας έχουν ε, φέρει το θέμα της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο. Υπήρξε μία έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ κλιματική αλλαγή ό,τι αφορά την αύξηση τη θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό και μα λέει αυτή η έκθεση ότι πρέπει να δράσουμε κατεπηγόντω και συλλογικά. Και σε αυτή τη χρονιά των, ε, που έχουμε, θα έχουμε ευρωεκλογέ, πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει ακόμα στην Ευρώπη. Βέβαια, μπορούμε να είμαστε αρκετά περήφανοι για τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Και η προεκλογική εκστρατεία του Κοινοβουλίου παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία να πούμε στου πολίτες μας τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και ε, να θέσει κάθε Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα τις θέσεις του για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε, αλλά ενδεχομένω να γνωρίζουν οι πολίτε μα, έχουμε υιοθετήσει ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο για το 2030, το οποίο καταφέραμε να πετύχουμε μόνο χάρη στην εξαιρετική ε, δουλειά, προσήλωση και αποφασιστικότητα των μελών του Κοινοβουλίου. Η Ενεργειακή Ένωση, λοιπόν, έχει πλέον θεσπιστεί. Ήταν μία από τι προτεραιότητε τη Επιτροπή Juncker, που υιοθετήσατε πριν από πέντε χρόνια. Η σωστή υλοποίηση ε, της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά το κλίμα και την καθαρή ενέργεια θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις ε, ε, εκπομπές ε, αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2030, πέραν του σημερινού στόχου του 40%, θα φτάσουμε κοντά στο 45% σε σχέση με το 1990. Αλλά μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Χάρη στο νομοθετικό πλαίσιο της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια που εθετήθηκε πρόσφατα, που θα δώσει έμφαση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση. Έχουμε ένα στόχο 32,5% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030 και μάλιστα αυτό θα αναθεωρηθεί προ τα πάνω το 2023. Αυτό δείχνει στους πολίτες μας ότι η κλιματική αλλαγή και τα ενεργειακά ζητήματα βρίσκονται ε, στην κορυφή της, ε, του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλουμε να, κάνουμε, να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το καλό παράδειγμα και ότι μετατρέπουμε τις δεσμεύσεις μας σε πράξεις. Όμως τώρα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον, προς το 2050. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις πολιτικές μας πέραν του 2030. Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ε, αυτό παρά μόνο αν μεταμορφώσουμε πραγματικά το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξής μας, ούτως ώστε να περάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα και στην ευημερία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό αυτό είναι και ο λόγο που η Επιτροπή υιοθέτησε τον Νοέμβριο μια ανακοίνωση για έναν καθαρό πλανήτη για όλου. Ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ε, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Και έτσι ανταποκριθήκαμε ε, στις ε, εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν με το όραμά της ε, θέλει να ε, προχωρήσει μπροστά με την κλιματική πολιτική. Έχουμε πέντε σενάρια τα οποία επιτυγχάνουν μία περικοπή κατά τουλάχιστον 80% μέχρι το 2050 με διάφορες ε, τεχνολογίες κυκλικότητα και ενεργειακή απόδοση. Για να είμαστε σαφεί, δεν επαρκούν αυτά για να φτάσουμε τον στόχο του 1,5 βαθμού. Και δεν είναι αυτή η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να φτάσουμε τον 1,5 βαθμό θα πρέπει να περιορίσουμε, ε, μάλλον να μηδενίσουμε τις εκπομπές ε, αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει δύο σενάρια που φτάνουν και επιτυχάνουν τον ε, στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Ένας βασίζεται στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, ο άλλος περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία συμπεριφορικής αλλαγής, κυκλοφορίας, κυκλικότητας μάλλον και άλλων μέτρων. Απαιτείται όμως ένας φιλόδοξος συνδυασμός τεχνολογίας και δράσης. Αυτό όχι μόνο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά και για να ξεχρονίσουμε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα βιώσιμο μέλλον, αύξηση των επενδύσεων σε ε, ανταγωνιστικές τεχνολογίες και για να προασπίσουμε ε, το βιωτικό επίπεδο των πολιτών μας. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε μια πιο αποδοτική οικονομία με λιγότερη εισαγόμενη ενέργεια ε, και μια οικονομία που παρέχει περισσότερες ε, θέσεις, ε, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Χαίρομαι που έχουν υιοθετηθεί ψηφίσματα στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Ελπίζω αυτό να γίνει και αύριο στην Ονομέλη. Είναι μεγάλη ευθύνη για εμά να δείξουμε ότι μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα όχι απλώ είναι δυνατή, αλλά ότι παρέχει και πολλέ οικονομικέ ευκαιρίε. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με του ε, πολίτε και την κοινωνία των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, επιτύχουμε μια κοινή κατανόηση ε, του μέλλοντο. Μαζί με την ομάδα μου έχω ξεκινήσει και έχω απευθύνει έκκληση προ όλε τι ευρωπαϊκές χώρες να ξεκινήσουν αυτό τον δημόσιο διάλογο και σας καλώ να συμβάλλετε κι εσείς στο όραμά μας για την Ευρώπη του 2050 και οι νέοι Ευρωπαίοι φυσικά εδώ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Είναι η ώρα να μιλήσουν. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε με τα μάτια μα τις επιπτώσεις κλιματική αλλαγή, αλλά οι περισσότεροι από εμά δεν θα είμαστε εδώ για να δούμε ε, πόσο δραματικά θα έχει αλλάξει ο πλανήτη το 2050. Οι νέοι Ευρωπαίοι που βγαίνουν τώρα στου δρόμου και όλο ένα και περισσότερο σε πολλέ πόλει σε όλη την Ευρώπη, θα είναι αυτοί που θα επομιστούν περισσότερο τι συνέπειε. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία μεταμόρφωσης ε, με μια μεγαλύτερη αίσθηση κατεπήγοντος από αυτή που έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να σταθεροποιήσουμε την κλιματική αλλαγή και να εκπληρώσουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Δεν έχει τελειώσει βέβαια ο χρόνος, αλλά πλέον δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και για δισταγμούς. Οι ενέργειες αλλά και τα λόγια αυτών των ε, νέων Ευρωπαίων είναι ένα σημαντικό έναυσμα για την ε, ε, προσπάθειά μας από εδώ και πέρα και οφείλουμε να αναλάβουμε δράση. Έχουμε δείξει πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί αυτό το μοντέλο ε, μπορεί να ε, αντιγραφεί και από άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο. Η κλιματική ουδετερότητα, λοιπόν, η οικονομική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Πρέπει λοιπόν, να ακούσουμε την πλειονότητα των Ευρωπαίων, ε, πρέπει να συμφωνήσουμε για το στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης, ευημερούσας και δίκαιης Ευρώπης το 2050. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Συνάδελφοι, θα περάσουμε στις πολιτικές ομάδες. Από το ΕΛΚ, τέσσερα λεπτά, ο κύριος Λίζα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Χέλμουτ Σμιτ, πρώην καγκελάριος ε, της Γερμανίας, είπε ότι όποιος έχει οράματα πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό. Στην πολιτική όμως χρειαζόμαστε οράματα και μάλιστα ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει παρουσιάσει ένα όραμα να είμαστε ουδέτεροι ως προς το κλίμα μέχρι το 2050. Και το καλό με το όραμα αυτό είναι ότι στηρίζεται από γεγονότα. Η δήλωση της Επιτροπής είναι σαφής. Μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη εάν επιδιώξουμε το στόχο αυτό σε όλη την Ευρώπη μαθητές ε, διαδηλώνουν ε, για το, για το κλίμα και εάν αύριο υιοθετήσουμε το ψήφισμα αυτό και στηρίξουμε το στόχο αυτό ενωμένοι, θα έχουμε πετύχει μια πρώτη επιτυχία. Φοβάμαι όμως ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν να ε, διαδηλώνουν και ελπίζω μάλιστα όχι σε ώρες ε, διδασκαλίας, ε, διότι δεν αποφασίζουμε μόνο εμείς και το Συμβούλιο πρέπει να υιοθετήσει την πρόταση αυτή και μάλλον θα είναι πολύ πιο δύσκολες εκεί οι διαπραγματεύσεις από ό,τι εδώ στο Κοινοβούλιο. Και για να παρακινήσουμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή και να αναλάβει συγκεκριμένα βήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι κάνουμε. Το ΕΛΚ βλέπει επικριτικά ε, τον στόχο του 55% μέχρι το 2030, διότι μόλις τώρα έχουμε υιοθετήσει πολιτική για το κλίμα και είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια προγραμματισμού. Φοβάμαι επίσης ότι τα κράτη μέλη που δεν θέλουν ιδιαιτερότητα προς το κλίμα στο Συμβούλιο θα έχουν επιχειρήματα που δεν θέλουμε να τους δώσουμε εάν υπερβάλλουμε στο ψήφισμα αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε βρει καλό συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ε, τον οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε αύριο. Για το ΕΛΚ είναι σημαντικό να έχουμε δίκαιη μετάβαση στην ε, ουδετερότητα, just transition. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ε, στις περιοχές που εξαρτώνται από την εξόριξη άνθρακα και θα πρέπει να ε, δώσουμε τη δυνατότητα στην βιομηχανία μας να παράγει χωρίς ε, να εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Για παράδειγμα, την ε, βιομηχανία χάλιβα. Στον τριμερή διάλογο, λοιπόν, θέλουμε να στηρίξουμε τις τεχνολογίες αυτές. Κυρίες και κύριοι, είδα τους ε, μαθητές που διαδηλώνουν ε, στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια. Είχα διάλογο μαζί τους. Έχουν τον πρώτο λόγο. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε απόγευμα και όχι κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας και σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση καλή και για τις επιχειρήσεις, διότι πολλές επιχειρήσεις μας λένε ότι δεν βγαίνουμε με την πρόταση αυτή. Δεν θα είμαστε υπόδειγμα εάν καταλήξουμε να είμαστε ουδέτεροι προς το κλίμα, αλλά έχουν μετικήσει όλες οι βιομηχανίες μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η αντίθεση θέσης απασχόλησης ή προστασία του κλίματος. Εμείς θέλουμε και τα δύο και γι' αυτό θέλουμε να υπερψηφιστεί το ψήφισμα αύριο χωρίς σημαντικές τροποποίησεις. Νομίζω ότι έτσι θα στείλουμε το σωστό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Λίζε. Από το SND 6 λεπτά ο κύριος Μπούλμαν. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, έχουμε προσκεκλημένους εδώ στο Κοινοβούλιο σήμερα 60 νέους ανθρώπους από 20 χώρες ε, στο, ε, στο θεωρείο και τους καλωσορίζουμε. Διότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και εκπροσωπούν ε, το ε, κίνημα η νεολαία για το κλίμα. Είναι πολύ θετικό λοιπόν ότι ε, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές μπορούν να συναντούν τους νέους στις εκλογικές του περιφέρειες. Σήμερα όμως έχετε την ευκαιρία να τους συναντήσετε εδώ πέρα κάτι ακόμα καλύτερο. Ε, πέρσι τον Αύγουστο η Γκρέτα Ντούνμπερκ ξεκίνησε το κίνημα αυτό η οποία αποφάσισε να διαδηλώσει μπροστά από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, κρατώντας ε, μία ταμπέλα που είχε ε, ζωγραφίσει μόνη της. Σήμερα όμως έχει γίνει κοινωνικό κίνημα, εκατοντάδες χιλιάδες σε πάνω από 70 χώρες, σε πάνω από 700 πόλεις διαδηλώνουν ε, με σύνθημα τις Παρασκευές για το μέλλον. Πρόκειται για κοινωνική επανάσταση η οποία έχει μεταφερθεί παντού. Και εμείς οι πολιτικοί, εμείς οι βουλευτές θα πρέπει να συμμετέχουμε στο κίνημα αυτό. Αυτή είναι απόλυτη υπεποίθησή πεποίθησή μου. Και ένα στοιχείο ακόμα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ στις θέσεις μας σήμερα. Ε, θα πρέπει να συνομιλήσουν μαζί μας, να μας πούνε ποια είναι τα αιτήματά τους, ε, να μας θέσουν ερωτήσεις και εμείς να τους απαντήσουμε. Και αυτή ήταν και η ιδέα κάποιων πολιτικών ομάδων, να τους καλέσουν να μιλήσουν σήμερα. Δυστυχώς όμως δεν πετύχαμε να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων για την πρόταση αυτό αυτή. Λυπάμαι πάρα πολύ που η συντηρητική, η φιλελεύθερη και η άκρα δεξιά μας στέρισε τη δυνατότητα αυτή για ανοιχτό διάλογο σήμερα. Δυστυχώς, εμπόδισαν να έχουμε ανοιχτή συζήτηση με τους νέους που κάθε εβδομάδα διαδηλώνουν στους δρόμους. Ίσως, ε, κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή στο μέλλον να τα καταφέρουμε καλύτερα. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι οι πολιτικές ομάδες που στήριξαν την πρόταση αυτή, τους προσκαλέσαμε στη συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων αυτή την ε, εβδομάδα. Και τους ρωτήσαμε τι επιθυμείτε. Και η απάντηση ήταν απόλυτα σαφής. Ήταν μια έκκληση για δράση. Είναι πάρα πολύ επίγον να κάνουμε κάτι. Παρακαλούμε μην αναβάλλετε. Παρακαλούμε μην δίνετε ευθυνές πολιτικές απαντήσεις. Παρακαλώ μην καθυστερείτε άλλο διότι αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ναι, έχουν δίκιο οι νέοι, διότι θέλουν να ζουν χωρίς φόβο, να έχουν προοπτική για το μέλλον τους, για τις μελλοντικές τους οικογένειες και θέλουν να ζήσουν χωρίς καταστροφές. Γι' αυτό θα ήθελα στους νέους ανθρώπους να πω ότι δεν αρκεί να χαμογελάμε, να κάνουμε σαν να ακούμε, χωρίς συνέπειες. Όχι. Πρέπει οι συνέπειες να είναι ριζικές εάν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη και εάν θέλουμε να φροντίσουμε όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη αυτόν να έχουν ένα μέλλον. Ε, εμείς λαμβάνουμε λοιπόν σοβαρά υπόψη μας το θέμα και έχω φροντίσει η πολιτική μου ομάδα να αναθεωρήσει το πολιτικό της πρόγραμμα. Και Είμαστε διατεθειμένοι να προσανατολίσουμε την πολιτική μας με τους, ε, ανάλογα με, τους στόχους βιωσιμότητας των Εθνών. Δεν επιτρέπεται όμως να υπάρχει και συζήτηση για το περιβάλλον χωρίς να λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική ασφάλεια στις κοινωνίες μας και να φροντίσουμε όλοι να κερδίσουν από την ε, εικόνα αυτή της μελλοντική κοινωνίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Η οικολογία δεν είναι κάτι για τους ε, λίγους και εκλεκτούς. Θα πρέπει να επενδύσουμε, να έχουμε μια σωστή περιφερειακή πολιτική, μια σωστή κοινωνική πολιτική. ο κύριος ε, Μακρόν ε, μαθαίνει σιγά σιγά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε δικαιοσύνη στις κοινωνίες μας. Δεν επιτρέπεται οι εργαζόμενοι μόνο να πρέπει να πληρώσουν ε, τη μεταρρύθμιση. Η οικολογική μεταρρύθμιση θα πετύχουμε μόνο εάν λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική μεταρρύθμιση. Και θα έχουμε κοινωνικό μέλλον εάν δημιουργήσουμε μια σωστή βιομηχανία και φροντίσουμε η... ο κόσμος αυτός να ζει σε ειρήνη με βάση τους φυσικούς πόρους. Άκουσα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άκουσα τον συνάδελφο Λίζε, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά. Φίλοι μου όμως, ε, εάν Όλοι έχουμε αποφασίσει τότε, ας τα κάνουμε αυτά στην νέα θητεία. Από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να δημιουργήσουμε ένα σύμφωνο βιωσιμότητας, ε, να έχουμε πολιτική βιωσιμότητας. Και να πω στους νέους, συνεχίστε να αγωνίζεστε, είμαστε, είμαστε στο πλευρό σας. Uh, Ευχαριστώ κύριε Μπούρμαν. Ως πρόεδρος θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε στην Ολομέλεια να κάνουμε μια ειδική ακρόαση στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία με νέους ανθρώπους για την κλιματική αλλαγή. Φαντάζομαι ότι πάρα πολύ θα υποστηρίξουν μια τέτοια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε εκ μέρου του ECR για 1,5 λεπτό η κυρία Βυσνιέσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Συμφωνία του Παρισιού ετοιμάζει ένα δρόμο για ένα καθαρό περιβάλλον. Χρειάζονται στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών. Δύσκολο καθήκον, αλλά μας δίνει και μια νέα προοπτική. Θα πρέπει να στοιχηματίσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για όλες αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες πρέπει να περάσουν από μετασχηματισμό, κυρίως εκείνες που βασίζονται στον άνθρακα, όπως η δική μου περιοχή, η Σιλικία. Ελπίζω οι σοσιαλιστές και το Άλντε να υποστηρίξουν το ψηφίσμα που μιλάει για μια δίκαιη μετάβαση που δεν αποκλεί κανένα, που δεν αποκλεί τα κράτη-μέλη που έχουν ένα ενεργειακό μείγμα δύσκολο όπου κυριαρχεί ο άνθρακας. Το... Στην Πολωνία, ας πούμε, βασιζόμαστε 180% στον άνθρακα, ενώ στη Γαλλία, ας πούμε, ε, το ενεργειακό τους μείγμα περιλαμβάνει μόνο κατά 2% άνθρακα. Εάν θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα καθαρό περιβάλλον, πρέπει να βοηθήσουμε εκείνες τις χώρες που βασίζονται στον άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν μια δίκαιη μετάβαση. Χρειάζεται υποστήριξη για τις ε, περιφέρειες αυτές που ζουν από τον άνθρακα. Αν δεν το κάνουμε, οι συζητήσεις μας θα είναι απλώς ε, μάτια χαμόγελα προς τους νέους. Ε, εγώ ξέρω ότι οι νέοι όμως είναι έξυπνοι. Ξέρω ότι θα συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει ο ενεργειακός αποκλεισμός. Αυτό σημαίνει φτώχεια. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε σήμερα διαδηλώσεις στους δρόμους του Παρισιού, ας πούμε, στη Γαλλία. Σας κάνω έκκληση, λοιπόν, υποστήριξη το ψηφισμά μου. Ε, ο κύριος Γκερμπράντι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή. Όχι μόνο επειδή η επόμενη γενιά βρίσκονται πρώτων πυλών, αλλά βρίσκονται και εδώ μάλιστα, στην αίθουσα αυτή, για να δουν κατά πόσο εμείς ε, προβλέπουμε για το μέλλον τους. Και ξεκαθαρίζουν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να καταστρέφουμε το δικό τους μέλλον. Έχουμε επίγνωση αυτού του γεγονότος και βρούμε αναλόγως. Πολύ φοβάμαι ότι η απάντηση είναι όχι όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και σε φορά γενικά τη συστηματική καταστροφή του περιβάλλοντο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πετύχει του στόχου που έχει θέσει για τη στρατηγική τη βιοποικιλότητας, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο έχουν υιοθετήσει μέτρα για να αντιστραφεί αυτή η τάση. Για το κλίμα. Πράγματι υπάρχει ε, θεσπισμένη νομοθεσία, πράγματι έχει αυξηθεί το ποσοστό του ευρωπαϊκού προπολογισμού που ε, αφορά την κλιματική αλλαγή. Φτάνει όμως αυτό. Όχι και το γνωρίζουμε όλοι πρέπει να υιοθετήσουμε και να, μάλλον να εκπληρώσουμε του στόχου που έχουμε θέσει για το 2030. Αυτό είναι σαφέ. Αλλά πρέπει να δράσουμε και σε όλου του άλλου τομεί πολιτική. Και τη Δευτέρα, πολύ φοβάμαι ότι αποδείξαμε για μια ακόμα φορά ότι απογοητεύουμε την ε, επόμενη γενιά. Βιώσ... Ψηφίσαμε για την βιώσιμη οικονομία. Και εξαιτία ε, τη δεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, καταψηφίστηκε οποιαδήποτε προσπάθεια φιλόδοξης ε, δράσης. Εμείς επικροτούμε τις πράσινες επενδύσεις, αλλά δεν έχουν καμία αξία αν δεν εξετάσουμε και όλες τις άλλες επενδύσεις. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Θα πετύχουμε λοιπόν μόνο αν όλες οι επενδύσεις είναι πράσινες. Πρόεδρε, σήμερα η επόμενη γενιά, η νέα γενιά, βρίσκεται εδώ, εκεί πάνω κάθονται. Λίγο χρόνο έχουμε στη θέσή μα. Σε μερικά χρόνια θα κάθονται εδώ, στα έδρανά μα. Και α αποφύγουμε το ενδεχόμενο εμείς να καθόμαστε εκεί πάνω και να κοιτάζουμε ντροπιασμένοι ε, το πόσο εκείνοι προσπαθούν να διορθώσουν τα δικά μας λάθη. Ευχαριστώ. Για τους ε, πρασίνους, ο κύριος Άικχαουτ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ και για την συζήτηση αυτή. Επιτέλου, πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση και πάλι την κλιματική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι πολλοί από αυτού που, έρχονται, που έρχονται σήμερα εδώ έχουν κουραστεί λίγο ε, να ακούνε, να του ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ε, δεν θέλουν ευχαριστίες, θέλουν δράση. Πριν από 10 χρόνια ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με ένα υπόβαθρο επιστημονικό στράφηκα προς την πολιτική, γιατί είδα ότι οι πολιτικοί δεν αναλαμβάνουν δράση και θεώρησα ότι πρέπει κάπως να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Και Πολύ λυπάμαι, Επίτροπε και εκπρόσωπε του ε, Συμβουλίου. Μιλήσατε για το 2050. Αν δείτε τις διαδηλώσεις ε, στο δρόμο, κανείς δεν μιλάει για ένα όραμα για το 2050. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Το αίτημα είναι θέλουμε δράση και τη θέλουμε τώρα. Πρέπει ως Ευρώπη να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξιών εδώ και τώρα. Και εσείς μιλάτε μόνο για ένα μακροπρόθεσμο όραμα και στρατηγική. Ο κύριος Λίζε μάλιστα λέει πρώτα να κάνουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μην μιλάτε και πολλά για τις ενέργειες και δράσεις, γιατί μπορεί αυτό κάπως να ταράξει ορισμένες χώρες. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Μιλούμε εδώ και μια κλιματική κρίση πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ένα από τα σλόγγαν λέει ότι αν το κλίμα ήταν τράπεζα θα τα είχαμε σώσει μέχρι τώρα. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αναλάβουμε δράση, να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό φαίνεται και από τις διαδηλώσεις που γίνονται στους δρόμους. Όχι μόνο ε, τα κινήματα των νέων. Αλλά ας πούμε την περασμένη εβδομάδα στο Άμστερνταμ 40.000 ε, άτομα, στις Βρυξέλλες 70.000 άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο και ζητούν δράση. Είναι ένα κοινωνικό, κοινωνικό κίνημα λοιπόν που δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε. Ζητούν από την Ευρώπη να κάνει περισσότερα. Και εφόσον μιλούμε για το μέλλον της Ευρώπης, αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η πράσινη απασχόληση. Ένα ακόμα σχόλιο προς τον συνάδελφο ε, Πίτερ Λίζε. Όταν μιλάτε για τις ε, μελλοντικέ θέσει εργασία, πρέπει και οφείλετε να μιλάτε για την ε, πράσινη μετάβαση. Άλλε περιοχές του πλανήτη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και επενδύουν. Δείτε την Καλιφόρνια. Αλλά ακόμα και την Ινδία με τις ηλιακέ επενδύσει, τι ηλεκτρικές μεταφορέ στην Κίνα. Εκείνοι σημειώνουν πρόοδο. Η δική σα αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει ε, στην ε, Κίνα, γιατί αυτές οι πολιτικές δεν εφαρμόζονται στη Γερμανία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα. Και να μην μιλήσουμε μόνο για στόχους. Θετικό είναι που κάποιοι ενοχλούνται, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μιας συζήτηση. Γιατί όλοι λένε ότι να, όλοι τα ίδια λέμε και έχουμε τους ίδιους στόχους, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν πάμε πέρα από τους στόχους βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα της, ε, ε, ε της ε, βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και τα προστατεύει η δεξιά σε αυτό το κοινοβούλιο. Κάποιοι για τη Γεωργία. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Γεωργία θα γίνει πράσινη, όπως και οι επενδύσεις και οι μεταφορές. και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση και την κλιματική διάσταση στις επενδύσεις μας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα και αύριο, αλλά και μετά με τις ευρωεκλογέ, που το διακύβημα θα είναι η ανάληψη δράσης. Όχι άλλα λόγια, μόνο πράξεις. Thank you. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ. μισή λεπτό από την Κούη, κυρία Βόιλαντ. Συνάδελφοι, η Κρέτα Τούνμπερκ δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι λέει την αλήθεια στην εξουσία. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι αποτυγχάνουμε όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, ε, δεν κάνουμε τα τολμηρά βήματα που πρέπει, δεν ε, βρισκόμαστε σε ηγετική θέση στο θέμα αυτό. Ε, πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ε, ανησυχούν πιο πολύ ε, για τις κοπάνες των νέων παρά για τις, τα μηνύματα των διαδηλώσεών τους. η, ο στόχος των δύο βαθμών Κελσίου δεν αρκεί πια. Ε, ε, μελέτη του IPCC μας έχει πει ότι πρέπει να περιοριστούμε στο 1,5 ε, βαθμό αν θέλουμε να αποτρέψουμε τις καταστροφές. Χρειάζεται λοιπόν γρήγορη και χωρίς προηγουμένου δράση. Είναι αυτό που απαιτείται, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε. Είναι σαν να βγάζουμε μια ομπρέλα για τον κατακλυσμό. Δεν αρκεί καθόλου σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και το θέμα εδώ δεν είναι ο πολιτικός συμβιβασμός, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε τα επιστημονικά στοιχεία. Αν ε, δεν στηρίξετε αύριο τις τροπολογίες ε, ζητώντας μείωση των εκπομπών κατά 50% είναι όχι μόνο προσβολή προς τους ακτιβιστές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από το θεωρείο αλλά τους λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον σας. Συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να πάρουμε ηγετική θέση στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Μπόιλαν. Από την ομάδα EFTD, ένα λεπτό, η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλες τις μεταφορές για το κλίμα. Τις ξέρουν οι πολίτες που βρίσκονται εκτός των θεσμικών οργάνων που διαδηλώνουν για να προστατεύσουν το μέλλον τους. Αλλά αυτό που περιγράφει καλύτερα ε, αυτό που ζούμε είναι ότι μαγειρεύουμε το πλανήτη σε χαμηλή φωτιά. Αυτή είναι η καλύτερη μεταφορά. Φυσικά υπάρχουν πολλαπλέ ευθύνε και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κάναμε αρκετά εμεί στην Ευρώπη. Κάναμε ό,τι έπρεπε για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον σε αυτόν τον πλανήτη, για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική μετάβαση ε, σε μια οικονομία με μηδενικέ εκπομπέ. Αλλάξαμε τον τρόπο παραγωγή μα και την κατανάλωση. Δεν νομίζω. Γιατί οι στόχοι που είχαμε μέχρι τώρα είναι απλώ επιχάρτου χάρτου και δεν αρκούν για να μειώσουν τη θερμοκρασία. Πρέπει να κάνουμε πράγματα από εδώ και πέρα. Κάνω μια έκκληση στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Ας ε, σταματήσετε την πολιτική λιτότητα, ας ε, σταματήσετε να περιορίζετε τι επενδύσεις ε, για την ενεργειακή μετάβαση. Α σταματήσουμε το ε, σύμφωνο σταθερότητα. Εγώ θα κατέβω στην πλατεία την Παρασκευή μαζί με όλου του νέου για να διαμαρτυρηθώ. Από το ΕΝΕΦ, e για ένα λεπτό, η κυρία Μελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα για όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο τρόπο το θέμα αυτό για να το αντιμετωπίσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα πρέπει επίσης ε, να συνειδητοποιήσουμε δύο φαινόμενα. Αυτό που αφορά την ανθρώπινη ευθύνη μετά από 200 χρόνια άγριας ε, βιομηχανικής ε, δραστηριότητας και ένα πάρτι με, τον, με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, επίσης, ε, τέσσερις βαθμοί αυξήθηκαν ε, η, θερμοκρασία στους πόλους ε, λόγω της μείωσης των, των στο, στο, βόρειο, στο βόρειο πόλο και εκεί δεν φταίει καθόλου η ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, ε, μη λέμε τα πράγματα όπως να είναι. Α σταματήσουμε τι ε, συμφωνίε ε, ελευθέρων συναλλαγών, α σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση, α κάνουμε σωστή διαχείριση, ε, ας αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής των αυτοκινήτων που μειώνει πάρα πολύ το κόστος τους κτλ. Ας βγούμε από τα δόγματα. Κυρία Μελά, ζητώ συγγνώμη. Εξατλήσατε το χρόνο σας. Και τώρα Τελειώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών και θα ζητήσω από τον Επίτροπο Κανιέντε να απαντήσει σε, αυτό, σε αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις παρεμβάσεις τους, τη φιλοδοξία τους και την ικανότητα να ακούν τους νέους. Θα μιλήσουμε στους νέου. Όταν μιλάμε για τους νέου, θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα ξεκάθαρα επί χάρτου. Το να λέμε ότι δεν, δεν έχει υπάρξει καθόλου δράση από πλευρά ε, κομισιών για την κλιματική αλλαγή δεν είναι σωστό. Δεν είναι αλήθεια. Αυτά τα πέντε χρόνια έγιναν πολύ περισσότερα για την κλιματική αλλαγή παραποτέ. Συμφωνήσαμε στο Παρίσι την πρώτη διεθνή δεσμευτική συνθήκη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικότατο εργαλείο για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Έχουμε μια συμφωνία που λέει ποιοι είναι οι στόχοι για να σταματήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή. Έχουμε την απαραίτητη νομοθεσία με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Έχουμε αυξήσει τη φιλοδοξία. Και ευχαριστώ όλου του Ευρωβουλευτέ από όλε τι πολιτικέ ομάδε που έχουν αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για τη βιώσιμη κινητικότητα, για μείωση των, του διοξιδίου του άνθρακα. Ε, κάνετε καλή δουλειά. Και η Κομισιόν λέει ότι το 2030 θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέες ρήτρε. Θα πρέπει να υπάρξει ε, δράση. Στους νέους θέλω να πω ότι θέλουν φιλοδοξία και ταχύτερη, ταχύτερη δράση. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν στην ανακοίνωση είναι ότι θα γίνουμε μέχρι το 2050 κλιματικά ουδέτεροι. Θα είμαστε δηλαδή ε, εμπρόθεσμοι. Δέκα χρόνια πριν α, χρειάζεται. Γιατί το IPPP λέει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί, δηλαδή η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2060. Εμείς θα το πετύχουμε 10 χρόνια πριν. Έχουμε νομοθεσία, έχουμε ρήτρε αναθεώρησης. Δεν είναι αρκετά αυτά. Φυσικά όχι. Και η, η επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο έχει τεράστιες ευθύνε. Και βλέπω ότι οι διάφοροι επικεφαλείς ψηφοδελτίων στι ομιλίε του μιλάνε για αυτό το θέμα. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει φιλοδοξία. Θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο και στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να υποστηριχθεί ο στόχο τη κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Έχουμε αυτό το στόχο. Φυσικά θα πρέπει να αυξήσουμε τη φιλοδοξία πιο πριν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θα γίνει τεράστια συζήτηση και στην προεκλογική εκστρατεία για το θέμα αυτό. Ακούνε οι νέοι. Η βιομηχανία ακούει, οι εργαζόμενοι ακούνε. Γιατί θα πρέπει να είναι μια δίκαιη κοινωνική μετάβαση αυτή. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή και να είναι όλοι άνεργοι. Αυτό δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε την εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών. Να αλλάξουν τη συμπεριφορά του, να δεχτούν την κινητικότητα με ηλεκτρικά οχήματα. Να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν του πόρου. Αυτό είναι μια επανάσταση. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που προτείνει η Κομισιόν είναι πάρα πολύ φιλόδοξα, αγγίζει όλους τους τομείς ε, της οικονομίας, απαιτεί διαρθωτικές αλλαγές. Θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλε τις πόλεις. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να απαντήσουμε στα αιτήματα και εκκλήσεις των νέων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να επικυρώσει φιλόδοξες ε, συμφωνίε, φιλόδοξου στόχου και θα πρέπει να υλοποιηθούν από την ε, επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο. Οι εργαζόμενοι των ορυχείων, το, της αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, όλοι οι εργαζόμενοι θέλουν μια δίκαιη κοινωνική μετάβαση. Θα πετύχουμε αν δεν αφήσουμε κανένα κατά μέρο, αν δεν αφήσουμε κανένα πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Υπουργό Τσότ, εξ του Συμβουλίου. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση, για τα σχόλιά σας και εγώ χαιρετίζω τους νέους που βρίσκονται στο θεωρείο σήμερα. Σημειώνω το γεγονό ότι εν γέννη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμμερίζονται πολλέ από τι φιλοδοξίε αλλά και επιφυλάξει ε, σε αυτό το θέμα είναι κέρια σημασία να σκεφτούμε πώς μπορούμε ε, να μεταμορφώσουμε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον για το περιβάλλον αλλά και για τους πολίτες, ε, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό βρίσκεται ε, σε ηγετική θέση σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Η Υπορουμανική Προεδρία, το Συμβούλιο, θα συνεχίσει το έργο ε, σε όλε τι πτυχέ του οράματο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να δώσουμε και να συμβάλλουμε κι εμείς όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα και θετικά στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Minister. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχω λάβει εννέα προτάσεις ψηφίσματο ψηφίσματος μετά από αυτή τη συζήτηση, μία από την Επιτροπή ε, Ήτρε, μία από την Επιτροπή Ένβη, μία από την ομάδα EFDD, μία από την ομάδα των Πρασίνων, από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, από την ομάδα των Φιλελευθέρων, πρόταση ψηφίσματος υπάρχει και από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και από την ομάδα του ΕΛΚ και από την ΚΟΕ. Σύνολο 9, λοιπόν. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Θα διακόψουμε για μερικά λεπτά. Θα ξεκινήσουμε στις 10 το επόμενο θέμα. Περιμένουμε τους συναδέλφους να καταφτάσουν. Ευχαριστώ και για την πειθαρχία σας. Ευχαριστώ και τους νέους ε, που βρέθηκαν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να ακούσατε ενθαρρυντικά πράγματα. Διακόπτουμε μέχρι τις 10.